Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Είστε έτοιμοι. Καθίστε παρακαλώ. Mm. Chers collègues, nous allons euh, commencer la séance de vote. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε τις προφορίες μας με την έκθεση Albrecht. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν έχω λάβει τροπολογία, δεν έχω λάβει πρόταση απόρριψης. Εγκρίνεται με βάση τη συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου η πράξη για την προστασία των φυσικών προσώπων ενάντια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κύριε Άλμπρεχτ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι ο θόρυβος στην αίθουσα είναι τέτοιος που καθιστά τη δουλειά μας σχεδόν αδύνατη. Πρόεδρε, η έγκριση της πράξης νομίζω συνιστά βήμα